Η πρόθεσή μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία ε, κατά το τρέχον έτος, κατά το 2012. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γεωργίευα. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση του θέματος. Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στι 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο τη ημέρας της άθεξης είναι η έκθεση του κύριου Νόιζερ. Σχετικά με τα συμβούλια τη Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Ελληνικής Πρόθεσης Καθολικής το 2030, θα ήθελα να δώσω στον εισηγητή το λόγο για 4 λεπτά. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση για την καθολική πρόσβαση στην ενέργεια είναι πολύ επίκαιρη στις αρχές του έτους 2012 γιατί τα Ηνωμένα Έθνη στην ε, Γενική Συνέλευση ε, κήρυξαν το έτος 2012 για διεθνές, ως διεθνές έτος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δύο είναι που για μένα και για όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν πάνω σε αυτή την έκθεση είναι σημαντικές. Η πρώτη έννοια είναι ότι θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η δεύτερη ότι θέλουμε μια καθολική πρόσβαση σε αυτές τις νέες μορφές ενέργειας. Γι' αυτό αυτές οι νέες πηγές ενέργειας θα πρέπει να είναι και οικονομικά εφικτές. Ε, εργαστήκαμε πάρα πολύ επικοδηματικά στην Επιτροπή Ανάπτυξης και με μη κυβερνικέ οργανώσει, παραδείγματο χάρη η Practical Action από το Λονδίνο και το Ιστιδικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντο τη Και η Γραμματεία μας ενίσχυσε για το πώς θα μπορούμε να προωθήσουμε την καθολική πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή τη στιγμή 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπων ζουν χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. 2,7 δισεκατομμύρια ε, μαγειρεύουν με βιομάζα σε τυχαίως ε, ε, φορείς. Το 20% του πληθυσμού της Κίνας έχει πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, μόνο το 5% όμως της, ε, ε, του πληθυσμού της υπαίθρου. Πρόσβαση σημαίνει και στη δυνατότητα να μαγειρεύει κανένας, να ζεσταίνεται. Η, πρό... η πρόσβαση στην ενέργεια δεν είναι ακόμα ένα στόχος της χιλιετίας ε, για την ανάπτυξη, αλλά χωρίς την πρόσβαση στην ενέργεια δεν μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι μας. Γι' αυτό προτείνουμε στην έκθεση αυτή στο νέο προσανατολισμό μετά το 2015 για τους στόχους ηλιετίας να αναφέρεται η πρόσβαση σε ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Σχολεία, εκπαίδευση, κέντρα υγειονομικά ή νοσοκομεία δύσκολα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς ηλεκτρισμό. Μα, μαγειρεύει κανένας και να στέλνεται με βιομάζα ε, σημαίνει πολλές φορές ε, εκατομμύρια θανάτους ανά έτος. Γι' αυτό πολλές χώρες ε, στην Αφρική απαγόρευσαν τη χρήση των, του ξυλοκάρβουνου για λόγους περιβάλλοντος ή υγείας. Βέβαια στην πράξη δεν μπορούν να το εφαρμόσουν κάτι τέτοιο και εξακολουθεί να παράγεται ξυλοκάρβονο. Χαιρετίζουμε λοιπόν για αυτή η Κομισιόν στη λεγόμενη Agenda for Change έχει συμπεριλάβει το θέμα των ασήμων πηγών ενέργειας και γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω τους κύριους στόχους της έκθεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη καλούνται να ε, υποστηρίξουν τους ε, στόχους του ΟΗΕ για την καθολική πρόσβαση μέχρι το 2030. Καλείται η Κομισιόν να συγκεντρώσει την σε μικρά σχέδια ανανεωσίμων ε, πηγών ενέργειας, γιατί μόνο έτσι μπορούν να έχουν επίδραση σε πολλούς ανθρώπους και αυτά θα πρέπει να διαδεθούν περισσότερα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλες σχετικές ευρωπαϊκές ε, τράπεζες δεν έχουν προσανατολιστεί σε μικρές ε, πήγες παραγωγής ενέργειας δεν επιτρέπεται. αυτό θα πρέπει να εκπροσωπούνται σημαντικά στη διαδικασία του Ρίο 2000. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους στόχους της ηλιατίας σαν ενεργησιακό στόχος οι ενώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ συνάδελφε Νόισερ. Περνάμε στη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΗ. Η συνάδελφος Βασέσκο έχει πρώτο λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στις ενεργειακές υπηρεσίες και αυτό πρόκειται να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο του κόσμου. Και αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό όσον αφορά τους φτωχότερους. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι η προσβασιμότητα στην ενέργεια θα πρέπει να αποτελέσει μια ε, ένα θέμα υψή τη προτεραιότητα όσον αφορά την ακριβή τη φτώχεια. Θα πρέπει επομένω να δούμε τι θα γίνει με τι σύγχρονε ενεργειακέ υπηρεσίε, κάτι το οποίο δυσκολεύει αυτή τη στιγμή ανηλίκου και γυναίκε. Επομένω, θα πρέπει στι τέντε κορυφή του Ιουνίου να συζητηθεί και αυτό και θα πρέπει να έχουμε ε, ίσως μια θεματική συνάντηση κορυφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα αυτά. Επίση, θα πρέπει να έχουμε επενδύσει από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα τη ενεργειακή υπηρεσία. Εγώ συμφωνώ με την πρόταση του να έχουμε χρηματοδοτικά προγράμματα για να ανανεώσιμες πηγές ε, ε, ενέργεια και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και στη χώρα μα γιατί θα έχουμε 300 εκατομμύρια που θα πάρουν η παραγωγή ενέργεια στην Ρουμανία. Ευχαριστώ, συνάδελφε Ο Κορέα Κάμπο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η πρόσβαση στις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας ε, πρέπει πραγματικά να συνιστά πρωταρχικό ευρωπαϊκό στόχο, ευρωπαϊκό στόχο, αλλά όχι μόνο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε καταπληκτικές τεχνολογικέ πρόοδου για τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από 20 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο για το 2015 έχουμε θέσει ως στόχο την καθολική πρόσβαση για τι ανανεώσιμε πηγές ενέργεια. Είναι λοιπόν πλέον αιτιολογημένο. Η υποσαχάρια Αφρική καταστρέφεται, μέρος της χλωρίδας καταστρέφεται λόγω της χρήσης της βιομάζας ως μοναδικό καύσιμο. Ε, γι' αυτό το λόγο πρέπει να επινοήσουμε νέες λύσεις. Στην Ευρώπη επίσης βασιζόμαστε υπερβολικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και θέλουμε ο καταναλωτή να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα. Τώρα αμφισβητείται όμω αυτή η αρχή από άλλου, κυρίω λόγω της ε, κρίσης που βιώνουμε ή λόγω των, ε, του λόμπινγκ που γίνεται υπέρ της πυρηνικής ενέργειας. Πρέπει λοιπόν να επινοήσουμε νέα μέτρα και νέες δράσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφο Ο συνάδελφος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, προσφάτως... Προσφάτως έλαβα μέρος σε ένα συμπόσιο που αφορούσε ενεργειακή πολιτική ε, και τις σχέσεις σε αυτό το πεδίο με τη ΕΠΑ. Εκείνοι τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα από εμά. Και αυτό διότι έχουν επεξεργαστεί ένα πάρα πολύ ισορροπημένο πρόγραμμα το οποίο ε, το υλοποίησαν. Εμεί δεν έχουμε πράξει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε εδώ πέρα είναι να έχουμε κάποιο είδου περισσότερη ποικιλία, περισσότερε εναλλακτικέ λύσει όσον αφορά του ενεργειακού πόρου. Άρα να κάτσουμε να δούμε τι εναλλακτικέ πηγέ συνέργεια υπάρχουν. Θα πρέπει να δούμε πώ είναι δυνατόν ίσω να χρησιμοποιήσουμε και με, με, με την γενετική επιστήμη τα βακτηρίδια. Αυτό, ξέρετε, το κάνουν οι Αμερικανοί και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν επομένως ε, την τεχνολογία για την παραγωγή δίζελ πετρελαίου. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την διασυνδεσιμότητα, τι θα πρέπει να γίνει με την ε, αποθήκευση ενεργεία, θέματα λέει, τα οποία, για μέτωπα στα οποία δεν τα πάμε καλά μέχρι τώρα. Ευχαριστώ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκα δεν έχει το μικρόφωνο τον άψει ακόμη. Ωραία, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νόιζερ. Υποστηρίζει μικρά αποκεντρωμένα προγράμματα για την παραγωγή ενέργειας σε αναπτυσσόμενες χώρες ενδιαφέρον και φιλόδοξο το πρόγραμμά του. Πλην όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει επαρκέ ικανότητε ούτω ώστε να προωθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δρομολογήσει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα τέτοιου είδου σε συνεργασία με άλλε βιομηχανοποιημένε και αναπτυσσόμενε χώρε, ούτω ώστε να έχουμε πολλαπλασιασμό των πόρων και μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα να βοηθήσουμε σε πολύ ευρύτερη κλίμακα αυτές τις χώρες σε σχέση με το που θα μπορούσε μόνη της να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, καταπολεμούν αυτό το σοβαρό πρόβλημα της ενεργειακής ένδιας ε, Δεν υπάρχει πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια για δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ε, πιστεύω ότι για τα αναπτυξιακά προβλήματα αυτό συνιστά προτεραιότητα. Η πρόσβαση λοιπόν στις πηγές ενέργειας ε, έχει καθοριστική σημασία κυρίω για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Αν δούμε όμω την κατάσταση που έχει εκεί παρατηρούμε ότι δεν έχει βελτιωθεί η πρόοδος ε, και τα νοικοκυριά δαπανούν μεγάλο μέρο των εισοδημάτων τους για κακή ποιότητα σε θέρμανση, για κακή ποιότητα σε καύσιμα. Για ποιο λόγο, διότι δεν έχουν καμία άλλη πρόσβαση και καμία ε, υποστήριξη από το κράτος. Χρειαζόμαστε καθαρές νέες πηγές ενέργειας. Γνωρίζουμε πώς μπορούμε ε, να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση ε, ενδέων κοινοτήτων σε αυτές τις πηγές ενέργειας. Χρειαζόμαστε κατά τη γνώμη μου ένα παγκόσμιο ταμείο που θα υποστηρίζει αυτά τα προγράμματα καθώς και τις επενδύσεις για την μείωση της παγκόσμιας ενδίας μέχρι το 2030 θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτή την καθολική πρόσβαση στην ενέργεια. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, συνάδελφο Μασερός. Συνάδελφος Τικάου. Σας ευχαριστώ πολύ. 84% του παγκοσμίου πληθυσμού ζουν στην Ήπεθρο και δεν έχουν πρόσβαση σε, σε ηλεκτρική ενέργεια. Πάνω από ένα 1.400.000 ε, ε, θανάτους έχουμε ε, από ατυχήματα που έχουν σχέση με το φυσικό αέριο. 3% των παγκοσμίων επενδύσεων όσον αφορά την ενεργειακή υποδομή θα γίνουν όσες επενδύσεις επομένως μέχρι το 2030 το οποίο θα αφορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο ώστε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμης πόρους ενεργείας, επομένως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα προγράμματα που έχουν, που έχουν, που έχουν προβλεφθεί με το 2015 και έτσι θα καταπονήσουμε και τη φτώχεια. Ευχαριστώ, Και Τικάου. Για να πρόγραμμα κατσάει η συνάδελφος Φρασικό Βαμπένοδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόσβαση στις σύγχρονες υπηρεσίες ενεργείας είναι μια προπόθεση για την εκκρίζωση τη φτώχεια. Διότι χωρί ε, μια τέτοια αρρύθμιση είναι καταδικασμένος ο κόσμος ζωή χωρίς αξιοπρέπεια, ζωή με, μεγάλη φτώχεια. Επομένως θα πρέπει ο τομέα να καταβάλει περισσότερη προσπάθεια, να επενδύσει περισσότερα όσον αφορά αυτή την ε, προσβασιμότητα. Όμως έχουμε πάρα πολύ λίγες αναπτυσσόμενες χώρες όπου υπάρχει ελπίδα για τέτοιου είδους προσβασιμότητα στην ε, ενέργεια. Οπότε χρειάζεται τώρα να υπάρξει περισσότερη οικονομική αρρωγή, που μέχρι σήμερα δεν ήταν αρκετή. Άρα θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας να, να προσπαθήσει περισσότερο ή στο μέλλον το, το, το, το μέσο πολιτικής ευρωπαικη Ένωσης θα είναι το μόνο ταμείο, το, η μόνη πηγή πόρων που θα υπάρχει ούτως ώστε να τονωθούν αυτές οι ε, επενδύσεις και έτσι να συμβάλλουμε στην εκκριση της φτώχειας. Όμως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό το μέσο πολιτικής θα υπάρχει στο μέλλον. Άρα θα πρέπει να, τελικά, να υπάρχει κάποιο είδους ε, ε, δέσμευση και έτσι να συνεχιστεί ε, η πολιτική αυτή. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέει κύριε Γεωργίευα, εξιότιμοι ε, κύριοι βουλευτέ, ε, εμεί θεωρούμε πάρα πολύ θετική την έκθεση που ε, μόλι τώρα συζητήσαμε και επίση όντω και εμεί θέλουμε να δεσμευτούμε ούτω ώστε οι στόχοι ενώ του 2030 θα πληρούνται και επίσης ενώ μας πηγές ενέργειας θα συστρατευτούν και αυτές θα επιστρατευτούν ούτως ώστε να πετύχουν αυτό το στόχο. Νομίζουμε ότι αυτό είναι όχημα για περισσότερη οικονομική ανάπτυξη και θεωρούμε ότι βοηθάται η υγεία, η παιδεία εκτός από την οικονομική ανάπτυξη. Καθαρή ενέργεια επίσης θα ωφελήσει, έτσι θα αντιμετωπίσουμε την μόνιση της ατμόσφαιρας και θα βοηθήσουμε σε καλύτερο επίπεδο δημόσιας υγείας ε, ε, όλα αυτά τα οποία προτείνετε εσείς είναι σύντομα τα δικά μας. Έχουμε και αυτή την ε, ατζέντα της αλλαγής. Αναγνωρίζετε πόσο σημαντική είναι η ομοιονάπτυξη, είναι η ενέργεια και εμείς κάνουμε τη φωνή της Ένωσης να ακουστεί στην ε, συνάντηση την παγκόσμια. Ο Επίτροπος ε, Πίμπαλτς επίσης καταβάλει προσπάθειες, ήρθε σε επαφή και με τον ε, Γενικό Γραμματέα Μπανκιμού σχετικά με αυτό. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία, ούτω ώστε να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένες συνθήκες που θα προλιάνουν το έδαφος για να πετύχουμε περισσότερα και να αντιμετωπίσουμε αυτές τι ε, προκλήσει που τελικά συμβαίνουν μία με την άλλη, δηλαδή και την κλιματική αλλαγή και την φτώχεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει δραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο ε, στις σχετικές ζυμώσει. οπότε βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους πρωταγωνιστές, αν όχι ο, ο βασικότερος πρωταγωνιστής σε αυτή την σκηνή. Τώρα, ο ρόλο μα είναι ενό δωρητή, μεγαλύτερο δωρητή, διότι 60% των πόρων που επιστατεύονται για αυτέ τι πολιτικέ προέρχονται από εμά. Και έχουμε την ε, Παγκοσμία Τράπεζα και έχω εργαστεί εκεί και μπορώ να σα ε, διαβεβαιώσω ότι όντω είναι πολύ φιλόδοξη η στόχη μα. Και επίση, μόνο οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χώρε που έχουν δεσμευθεί για τέτοιου ε, στόχου που αφορούν τι ανεσμευτικέ ενέργειε, Έχουμε το Ρίο συν 20 που είναι μια ευκαιρία μοναδική. Πρόκειται να μα βοηθήσει να ε, επιστρατεύσουμε ε, νέε πολιτικέ και επομένω να μπορέσουμε να έχουμε και του αναγκαίους σχηματικού πόρου, Έχετε παίξει και εσείς σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί ούτως ώστε να υποστηριχθούν ε, αυτοί οι στόχοι που συζητήσαμε. Θα πρέπει να έχουν προστασιμότητα οι φτωχοί. Πήγα στο Τσάζ, στην Ιγυρία και σε άλλε φτωχές χώρε και είδα από κοντά τι γίνεται. Θα πρέπει ομένως και εμείς να προσπαθήσουμε πάρα πολύ όσον αφορά τι ε, ε, νέε ενέργεια, γιατί θα πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο, το φτωχό, να έχει προσβασιμότητα ε, στο καθαρό νερό. Επομένως βλέπουμε το πόσο σημαντική είναι αυτή η στόχη και να πετύχουμε κάποιες μη κεντροκατευθυνόμενες και αποκεντρωμένες λύσεις. Ε, πέραν της ανακοίνωσης θα πρέπει να βοηθήσουμε να έχουμε νέες πηγές ενέργειας για όλους και βιώσιμες. Όλοι να έχουν προσβασιμότητα με βιώσιμο τρόπο εις αυτές τις πηγές ενέργειας. Οπότε θα πρέπει να δούμε με ποιο μηχανισμό οι αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορέσουν να προσχωρήσουν σε προγράμματα μέσω των οποίων θα έχουν την κατάλληλη αρρωγή παντός για αυτή την στρατηγική της προσβασιμότητας δέσμευση από τους ε, εταίρους μας. Και έτσι να πραγματοποιήσουμε το στόχο της, ε, του να έχουν περισσότερες επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Σας ευχαριστώ που μας στηρίξατε και συγκεκριμένα την Επιτροπή Ανάπτυξης που πάντοτε είναι στο πλάι μας. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, ε, Επίτροπε κύριε Γεωργίευα. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση του θέματο αυτού. Η ψηφορία θα γίνει σήμερα στι 12 το μεσημέρι. Επόμενο σήμερα σήμερα στη διάλεξη. Έκθεση του συναδέλφου Σμιτ για την ετήσια έκθεση για την φορολογία. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εισηγητή για 4 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητή Επίτροπε. Χαίρομαι πάρα πολύ